Przewodniczący! Wznawiam posiedzenie. Αγαπητοί συνάδελφοι, επαναρχίζει η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να καλωσορίσω στην αίθουσα της Ολομέλειας τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου καθώς και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε ενώπιον μας τον πρόεδρο της ε, Κομισιόν καθώς και τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Σουηδίας. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εγκρίνετε τα κείμενα της χθεσινής συνεδρίασης και τα πρακτικά. Έχετε κάποιες παρατηρήσεις σχετικά σε σχέση με τα πρακτικά ή τα εγκεκριμένα κείμενα. Εάν δεν υπάρχει καμία ε, αντίρρηση θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί. Ο κύριος Σούλτς όμως θα ήθελε το λόγο. Έχετε το λόγο κύριε Σούλτς. Χωρίς μικρόφωνο κύριο Σούλτς. Δεν έχω κάποια ε, παρατήρηση για τα πρακτικά, αλλά θέλω να αναφερθώ σε ένα επεισόδιο που έλαβε χώρα στην σημερινή συνεδρία στην πρωινή. Ο κύριος Κίνγκερ Γκάρτς από την δική μου, η κυρία Κίνγκερ Γκάρτς μάλλον, πρώην υπουργό της Ουγγαρίας, α, αντιμετωπίστηκε από την κυρία ε, Γιώβικ Μόρετς από το φασιστικό κόμμα Γιώβιτς με τρόπο ο οποίος είναι απόλυτα απαράδεκτος. Η συνάδελφός μας έχει αγωνιστεί για να υπάρξει πραγματικά μια δημοκρατική συνέχεια στην Ουγγαρία και μια πραγματικά σωστή αντιμετώπιση μετά από τα κομμουνιστικά καθεστώτα. Λοιπόν, ζητώ από την εκπρόσωπο του Φασιστικού Κόμματος να αποσύρει τα σχόλιά της. Λέει και ο πρόεδρο, κύριε Σούλτ, για τη δήλωσή σα. Η κυρία Γκιούντς ζήτησε το λόγο επίσης και για ένα προσωπικό θέμα. Η κυρία Γκιούντς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να λάβω το λόγο. Εγώ λυπούμε για το γεγονός ότι ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αναφέρεται αυτό το γεγονός το οποίο αναφέρθηκε. Το κόμμα το οποίο αναφέρθηκε εδώ έχει μια στρατιωτικού χαρακτήρα οργάνωση και καταπιέζει Εβραίους, Τσιγκάνους και άλλες μορφές μειονότητας. Το κόμμα αυτό λοιπόν έχει αυτή τη μορφή στην Ουγγαρία. Ακόμα και ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει έρθει εδώ με την ε, στολή αυτού του κόμματος. Είναι ένα ξενοφοβικό κόμμα, ένα κόμμα ομοφοβικό, ένα κόμμα κατά των τσιγκάνων και έχει αντιμετωπίσει με ένα τρόπο την Ουγγαρία σαν να είναι, όπως λέει, απικία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άκρες δεξιές στην ε, Ουγγαρία έχουν διοργανώσει πολλές ε, ε, διαδηλώσεις, έχουν τραυματίσει <clears throat> αστυνομικούς, έχουν προξενήσει ζημίες στο, στο κτίριο της Ουγγρικής τηλεόρασης έχουν προσπαθήσει να διαταράξουν τον εορτασμό της εθνικής εορτής της Ουγγαρίας. Επομένως, η αστυνομία δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει στην Ουγγαρία όλες αυτές τις εξτρεμιστικές δυνάμεις. Και είναι φανερό για όλους ότι υπάρχουν πραγματικά προβλήματα με αυτές τις εξτρεμιστικές οργανώσεις και όχι με τον τρόπο με τον οποίο τις έχει αντιμετωπίσει η αστυνομία. Θέλω λοιπόν να τονίσω όταν η Ουγγαρία ήδη στο εσωτερικό της έχει να αντιμετωπίσει δυνάμεις οι οποίες αντιμετωπίζονται σαν να μην είναι δημοκρατικές, τότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό όταν γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν μπορεί να ομιλεί λοιπόν κύριε Μωράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Μπόλτον και μετά πιστεύω ότι μπορούμε να σταματήσουμε τις προσωπικές δηλώσεις από την πλευρά των βουλευτών. Κύριε Μπόλτον. Βάσει του κανονισμού, Πρόεδρε, ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Σούλτς να μας πει πώς ε, παίρνει το θάρρος να πάρει το λόγο και να χαρακτηρίσει φασιστικό ένα τέτοιο κόμμα. Ένα κόμμα που έχει τόσο καθοριστικό ρόλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 431.000 Ούγγροι πολίτες ψήφισαν υπέρ του κόμματος αυτό. Πώς μπορείτε να τους χαρακτηρίζετε φασίστες. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτόν τον τόνο τις προσωπικές τοποθετήσεις. Την Τετάρτη θα προσυπογράψουμε 22 αποφάσεις ε, συναπόφασης βάσει και του άρθρου 74 του κανονισμού. Και στις 15 του μήνα θα έχουμε και την υπογραφή για τον δημοσιονομικό κανονισμό. Και όλα αυτά βάσει τη ε, χθεσινής